συστήματος EU-10 που πραγματικά θα είναι αποτελεσματικό. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα από τα μειονεκτήματα και ελπίζω να το λάβετε υπόψη σα κατά την εκτέλεση των επόμενων βημάτων από εδώ και πέρα. Ε...